Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Κυρίσω την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής μας και καλωσορίζω θερμά την κυρία Μακάβεν, η οποία είναι πρόεδρος της Επιτροπής Αναπτυξιακής. Έχουμε μια σημαντική ανακοίνωση για ένα ταμείο που πρέπει ε, να παρατείνουμε τη διάρκεια του. Στο μεταξύ, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Να ξέρετε ότι το σημείο 7 αναβάλλεται. Πρόκειται για την έκθεση που εγώ θα σας παρουσίαζα για το ψήφισμα του Συμβουλίου που έχει να κάνει με το Brexit. Ε, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι για το θέμα αυτό περιμένουμε στο ακουστικό μας. Λοιπόν, δύο λόγια τώρα να σας ενημερώσω για την άτυπη συνάντηση που είχαμε τους Υπουργούς Εξωτερικών Γενικών Υποθέσεων της 12ης Μαρτίου στο Βουκουρέστι. Η διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και για τους ίδιους πόρους εκλήθη στις 12 Μαρτίου στο Βουκαρέστι, προσκαλέστηκε να συμμετάσχει σε μια άτυπη συνάντηση με τους υπουργούς των 28 ετών ε, κρατών χωρών σχετικά με το άτυπο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Εκεί θέλαμε να στηρίξουμε τις ε, κύριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο 2021 με 2027. Ε, για πρώτη φορά να έχουμε συνάντηση απευθείας με όλους τους υπουργούς και υφυπουργούς που εδρεύουν στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων αντί να έχουμε ενδιάμεσους με την Προεδρία του Συμβουλίου. Έτσι λοιπόν ε, μπορέσαμε να εξηγήσουμε ποιες είναι δικές μας ε, προτιμήσεις για τη διαδικασία διαπραγματεύσεων όσον αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τα ε, τομεακά προγράμματα, τους ίδιους πόρους, τα όρια, την ευελιξία, τις οριζόντιες αρχές και την αναθεώρηση στα μισά του δρόμου. Ε, παρόλο που είχαμε περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή μα, η ανταλλαγή απόψεων που είχαμε με του υπουργού ήταν ειλικρινή και πιστεύω και ποιότητα. Κάποιοι υπουργοί στήριξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην προσπάθειά του να πετύχει νέους ιδίους πόρου και να προβλέψει πραγματικούς μηχανισμούς ευέλικτους πέρα από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και να μπορέσει έτσι να προστατεύσει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίπτωση που δεν λειτουργεί καλά το κράτος δικαίου σε κάποια χώρα. Ε, όπως βέβαια περιμένουμε, κάποιοι από τους καθαρούς ε, συνεισφορείς ε, εκφράστηκαν υπέρ ενός ε, χαμηλού προπολογισμού 1% το πολύ και χωρίς άλλους ίδιους πόρους. Είχαμε την εντύπωση ότι το Συμβούλιο δεν είχε προχωρήσει και πολύ στις δικές του εργασίες και ότι θα είναι δύσκολο να πετύχει το στόχο που έχει το ίδιο καθορίσει, δηλαδή να καταλήξει σε θέση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το φθινόπωρο του 2019. Εγώ από τη δικιά μου την πλευρά ζήτησα από τους Υπουργούς να καθορίσουν τη δικιά τους στρατηγική άποψη όσον αφορά το ρόλο και τις αρμοδιότητες της Ευρώπης να εκφραστούν και να εντοπίσουν τα κοινά αγαθά και ποιοι θα πρέπει να είναι οι πόροι που θα πηγαίνουν από το εθνικό επίπεδο στο ευρωπαϊκό. Του ζήτησα να προσπαθήσουν να σκεφτούν πέρα από τα συνηθισμένα. Τους είπα out of the negotiating box. Να σκεφτούν κάπως ασυνήθιστα. Δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Less of the same. Οι διοργανικές επίσης επαφές πρέπει να ενισχυθούν. Αυτό είναι κάτι το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει εδώ και πολλού μήνε. Κάποια θέματα θα συζητηθούν από τους διαπραγματευτέ μας μετά τις εκλογές και θα κληθούν στο επόμενο άτυπο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που θα γίνει υπό Φιλανδική Προεδρία αυτή τη φορά. Να πω και δύο λόγια τώρα για τη συνάντηση που είχαμε με τον Επίτροπο Έτιγκερ. Συναντήθηκα με τον Επίτροπο στο Στρασβούργο και συζητήσαμε για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο αλλά και για του ίδιου πόρου, Και ο επίτροπο ήθελε να μα ενημερώσει για διάφορα πράγματα που μάλιστα είναι και εκτό πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Όσον αφορά αυτό, ο επίτροπο ήθελε να εκφράσει την εμπιστοσύνη του λέγοντα ότι θέλουν συμφωνία οι χώρε μέλη ήδη τον Οκτώβριο του 2019. Όπω είπα και πριν από λίγο, εμεί δεν σχηματίσαμε αυτή την άποψη όταν συναντηθήκαμε με του υπουργού στο Βουκουρέστι όμω. Τώρα όσον αφορά το Brexit, ο Επίτροπος επέστησε την προσοχή μας στο χάσμα χρηματοδότησης το οποίο απορρέει εφόσον έχουμε ένα Brexit χωρίς συμφωνία και χωρίς μεταβατική συμφωνία δηλαδή με 6 δισεκατομμύρια για το 2019 και 12 δισεκατομμύρια για το 2020. Αυτό θα είναι το χάσμα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ο Επίτροπος προβλέπει ένα διορθωτικό προπολογισμό για το 2019 που προβλέπει αύξηση των συνεισφορών των 27 χωρών μελών και από την άλλη μεριά και μία ε, μείωση των δαπανών. Εγώ αρχίζω να αναρωτιέμαι πάντως και να σκέφτομαι ότι ίσως τελικά το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως. Κάτι το οποίο θα αποδεικνύει και την ε, αντοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα όσον αφορά τον προπολογισμό για την Ευρωζώνη, ο Επίτροπος περιέγραψε ένα διχασμένο συμβούλιο, ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές ομάδες χωρών και ίσως να έχουμε μία πρόταση τον Ιούνιο. Ο Επίτροπος λοιπόν δίνει την εντύπωση ότι ασκεί πίεση στο Κοινοβούλιο έχει υπογράψει με τη Ρουμανική Προεδρία επιστολή, η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, με την οποία καλεί όλες τις επιτροπές να ψηφίσουν πριν από την Ολομέλεια του Απριλίου, που είναι και η τελευταία της θητείας αυτής. Κάτι το οποίο βέβαια οδήγησε σε αντιδράσεις και σε διαμαρτυρίες, γιατί εάν ο Επίτροπος πρέπει να πιέσει, τότε πρώτα απ' όλα πρέπει να πιέσει το Συμβούλιο. Γιατί εμεί είμαστε έτοιμοι από τον Νοέμβριο για διαπραγματεύσει, αγαπητοί συνάδελφοι. Και επειδή βλέπει ο επίτροπο ότι δεν υπάρχουν θετικέ αντιδράσει, τι κάνει? Ε, συγκαλεί τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους εισηγητές να έχουν νέα συνεδρίαση προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία. Και αναρωτιέμαι κατά πόσο είναι αυτός ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε, αγαπητοί συνάδελφοι, γνώμη μου είναι ότι πρέπει να ενημερώσουμε τον Επίτροπο και να του πούμε ότι δεν πρέπει να μας πιέζει και να καταπιέζει τα δικά μας τα προνόμια. Οι δύο βραχίονες του προπολογισμού είναι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Και η Επιτροπή παίζει το ρόλο του διαμεσολαβητή. Οπότε ο Επίτροπος μπορεί να θέλει πριν από τα τέλη Οκτωβρίου να τα έχει λύσει όλα, αλλά δεδομένο των προθεσμιών και της έλλειψης προετοιμασίας στο Συμβούλιο, δεν το βλέπω. Από ό,τι είδαμε εμεί στο Βουκουρέστι, από ό,τι φαίνεται, όλοι περιμένουν ότι κάποια στιγμή οι επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων θα συνεδριάσουν και θα ε, συμφωνήσουν για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, κρίνοντας ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες το Κοινοβούλιο, όποιο και αν είναι το περιεχόμενο του εγγράφου, θα δώσει τις ευλογίες του και ότι τα υπόλοιπα θα μείνουν για την επόμενη θητεία. Τώρα, οι αποφάσεις των συντονιστών, άλλο θέμα, που σας έχουν ανακοινωθεί από τα πρακτικά της 7ης Μαρτίου. Τα έχετε στους φακέλους σας φαντάζομαι. Οπότε, μπορώ να θεωρήσω ότι εγκρίνονται. Και επίση υπάρχουν και τα πρακτικά τη συνεδριάσεώ μα τη 14η και 26η Φεβρουαρίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, τότε θεωρούνται τα πρακτικά αυτά εγκεκριμένα. Δεν βλέπω αντιρρήσει. Εγκρίνονται λοιπόν. Οπότε το σημείο στο οποίο θα περάσουμε τώρα είναι το καταπιστευματικό ταμείο Trust Fund για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Πρόκειται για το Ταμείο Μπέκου. Είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζουμε από κοινού με την Επιτροπή Ανάπτυξης. Οπότε χαιρετίζω και πάλι εδώ την παρουσία της κυρίας Μακάβεν και του συναδέλφους της Επιτροπής ανάπτυξη. Έχει ζητηθεί παράταση για ένα ταμείο το οποίο δημιουργήθηκε για μία πενταετία και που εκπνέει στι 30 Ιουνίου του 2019 και εμείς πρέπει να αποφασίσουμε για μια παράταση των 18 επόμενων μηνών. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στη Λίντα Μακάβεν πρώτα απ' όλα για να μας εισαγάγει σε αυτό το θέμα. Σε ευχαριστώ αγαπητέ Ζαν. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να έχουμε μια κοινή συνεδρίαση σχετικά με το Ταμείο Μπεκού. Πριν πάρω το λόγο όμως για το Ταμείο αυτό, θα ήθελα να καλωσορίσω μία ομάδα επισκεπτών από τη Νέα Καλλιδονία που βρίσκονται εδώ κατόπιν πρόσκληση ε, του Αντιπροέδρου του κ. Μπόγκα της Επιτροπής ανάπτυξη, που δυστυχώ δεν μπορεί να είναι παρόν ο ίδιο. Είστε εδώ. <laughs> Καλώς ήρθατε. Γνωρίζω ότι για πολλού είναι η πρώτη σα επίσκεψη εδώ στι Βρυξέλλε, για πολλού μάλιστα η πρώτη σα επίσκεψη στην Ευρώπη. Σα ε, καλωσορίζουμε θερμά. Σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ. Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε στο Brexit και ότι αναμένουμε τις εξελίξεις. Ε, όλοι βρισκόμαστε εδώ εν αναμονή των εξελίξεων στο Λονδίνο, διότι όπως έχουν τα πράγματα δεν γνωρίζω εάν θα είναι η τελευταία συνεδρίαση της ΔΕΒΕ στην οποία θα προεδρεύω, αν θα είναι η τελευταία μου εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Ε, ε, βρισκόμαστε λοιπόν γενικά εν αναμονή Η συνεδρίασή μα ε, είναι κοινή με την Επιτροπή Ανάπτυξης. Πολλοί συνάδελφοι όμω δεν είναι παρόντες, διότι έπρεπε να βρίσκονται στην κοινή κοινοβουλευτική συνέλευση στο Βουκουρέστι. Δεν καταφέραμε να βρούμε άλλη κοινή ημέρα των δύο ε, επιτροπών μα ε, πριν τι εκλογέ και όπω είπατε πρέπει να λύσουμε το θέμα τη παράταση του Ταμείου πριν τι εκλογέ, διότι το Ταμείο όπως έχει λίγη τον ε, Ιούνιο. Γιατί συζητάμε λοιπόν ε, το Ταμείο αυτό λόγω της αλλαγής των κανόνων στον δημοσιονομικό κανονισμό. αγωνιστήκαμε ώστε να έχει το Κοινοβούλιο ε, ενισχυμένο λόγο ε, και πράγματι έχει τώρα όσον αφορά το Ταμείο αυτό, τα θεματικά ταμεία και όσον αφορά την παράταση των ε, καταπιστευματικών ταμείων. Ωστόσο, επειδή είναι νέος κανόνας, δεν έχουμε στον εσωτερικό μας κανονισμό σαφή διαδικασία. Η Επιτροπή επιτροπές μας ε, ε, προϋπολογισμών ε, ανάπτυξης και διεθνούς εμπορίου είναι οι τρεις αρμόδιες επιτροπές. Είναι λοιπόν αυτή η διαδικασία που θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή αλλά συνομιλήσαμε και με τον πρόεδρο της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, ώστε το μελλοντικό κοινοβούλιο, η επόμενη θητεία, να καθορίσει μια διαδικασία. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή μια διαδικασία, θα πρέπει όμως να έχουμε μια επίσημη διαδικασία στην επόμενη θητεία. Θα ακούσουμε σύντομα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την παράταση του Ταμείου. Θα μας πει η Επιτροπή γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι απαραίτητο και μετά από τη σημερινή μας συζήτηση οι συντονιστέ των δύο επιτροπών μας με γραπτή διαδικασία θα αποφασίσουν σχετικά με την παράταση. Η διαδικασία αυτή θα έχει τη μορφή επιστολή προς τον πρόεδρο Ταγιάννη, όπου θα του ζητείτε να ενημερώσει την Ολομέλεια ε, για την αποφασή μας, καθώς και ε, τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής γραπτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας ε, πει λοιπόν κάποια στοιχεία, να δώσω όμως εγώ γενικά το πλαίσιο. Ήταν το πρώτο καταπιστευματικό ταμείο και στόχος ήταν να συγκεντρώσουμε τη, τους πόρους ε, για την κεντροαφρικανική δημοκρατία μετά από την κρίση στην οποία έπεσε η χώρα το 2012-2013. Πέρα από κάποιες ε, δωρεές 133 εκατομμυρίων από το EDF και από τον ε, Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Ε, κάποια άλλα κράτη-μέλη ε, συνεισφέρουν, όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελβετία και η Ολλανδία. Αυτή τη στιγμή σε 239,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό του Ταμείου. Θα μιλήσω σε λίγα λεπτά για το θέμα αυτό, διότι πήγα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και είδα τον αντίκτυπο του Ταμείου αυτού. Η λέξη «μπέκου» στη γλώσσα σάγκο της χώρας σημαίνει ελπίδα. Και πράγματι τα όσα είδα φαίνεται ότι φέρνουν ελπίδα στους ανθρώπους που ζουν υπό φρικτές συνθήκες. Συμμετείχα σε συνάντηση του Συμβουλίου του ε, Ταμείου, διότι είμαστε παρατηρητές εμείς στο Κοινοβούλιο, ε, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στις 30 ε, Νοεμβρίου συμμετείχα λοιπόν στη συνάντηση αυτή και συστήθηκε παράταση του Ταμείου μέχρι το 2020 και γι' αυτό έχουμε τη διαδικασία αυτή σήμερα. Η Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία είναι η πιο φτωχή χώρα στον κόσμο σύμφωνα με τον δίκτυο ανθρώπινης ανάπτυξης. Ε, είναι μια χώρα υπηρετική, χωρίς παράλια. Ε, υπάρχει μακρά ιστορία ε, αμέλειας και έλλειψης κοινωνικών υπηρεσιών. Πέρσι, όταν επισκεφτήκαμε τη χώρα, διαπιστώσαμε ότι η κατάσταση ως προς την ασφάλεια είναι πολύ δύσκολη στη χώρα αυτή. Το ταμείο αυτό, αυτό που μπορεί να κάνει σε σχέση με άλλα ταμεία είναι γρήγορα να συγκεντρώσει χρήματα για συγκεκριμένα έργα. Είδαμε λοιπόν συγκεκριμένα έργα, πολύ μικρά, ε, για να βοηθήσουν γυναίκες να δημιουργήσουν μικρές επιχειρήσεις ε, στην πρωτεύουσα. Την πρωτεύουσα Μπανγκή. Είδαμε και κάποια άλλα προγράμματα. Είναι μια χώρα όπου υπήρχαν πολλές ε, κοινοτικές εντάσεις ε, πολλοί άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και γίνονται προσπάθειες να επανέλθουν οι άνθρωποι αυτοί στα σπίτια τους, ε, να οικοδομηθούν νέα σπίτια και να στηριχθούν οι κοινότητες. Ε, ο συνάδελφός μου Νόρβερτ Νόιζερ. Οι δύο συντονιστές του ΕΛΚ και του Κοινοβουλίου δυστυχώ δεν μπορούν να είναι παρόντες εδώ σήμερα. Με συνόδεψαν όμως. Μετά την δική μας επίσκεψη το 2017 η κατάσταση επιδεινώθηκε. Φέτος τον Φεβρουάριο όμως υπεγράφει η Συμφωνία Ειρήνευσης ανάμεσα στις διάφορες φατρίες, διότι χωρίς ειρήνη στη χώρα αυτή είναι πολύ δύσκολο να δούμε πώς θα μπορέσει να υπάρξει ανάπτυξη. Πολλά χρήματα έχουν δαπανηθεί για να εκπαιδευτεί ο στρατό. Εμεί, όταν βρισκόμασταν εκεί, ε, δεν μπορούσαμε να εγκαταλείψουμε την πρωτεύουσα. Δεν ήταν ασφαλέ να εγκαταλείψει κανεί την πρωτεύουσα. Νομίζω ότι τώρα έχουν υπάρξει κάποιε βελτιώσει ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βοηθήσει τον στρατό να εκπαιδευτεί για να ξαναλάβει ε, τον έλεγχο της χώρας αυτής. Πάντως είχαμε ούτως ή άλλως τη Συμφωνία Ειρήνευσης αυτή του Φεβρουαρίου ε, θα ήθελα να καλέσω τον συνάδελφο από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ να μας μιλήσει για την παράταση του Ταμείου και να μας ενημερώσει σχετικά με την κατάσταση. Φρανσέσκο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, λέει η κυρία Φραντσέσκα Ντιμάουρο, ευχαριστώ για τη συνεδρίαση αυτή. Με μεγάλη χαρά ήρθαμε εδώ. Ε, υπάρχει ένα θαυμάσιος ε, υπερασπιστής αυτού του ταμείου. Ήρθατε, πήγατε επί τόπου και είδατε τι μπορεί να καταφέρει αυτό το ταμείο. Κάνετε και μία εισαγωγή για το ίδιο το καταπίστευμα. Δεν θα επαναλάβω όλα αυτά τα πράγματα. Δημιουργήθηκε το 2014 ε, για να αντιμετωπιστεί η κρίση σε μια χώρα η οποία ήταν σε αβυσαλαία κατάσταση. Ε, η παρουσία του ίδιου του κράτους ήταν ανύπαρκτη μάλλον. Είπαμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη νέα ευκαιρία που έχουμε με τα καταπιστεύματα για να παρεύουμε σε μια χώρα όπου δεν υπάρχει κυβέρνηση, όπου ο λαός έχει εκτοπιστεί σε μεγάλο βαθμό, υπάρχουν τεράστιες ανθρωπιστικές ανάγκες και υπήρχε βέβαια ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά θέλαμε να μην εστιάζουμε μόνο στο ανθρωπιστικό κομμάτι, αλλά να στηρίξουμε λιγάκι και τις μικρές δομές που, και τη μικρή διοίκηση που υπάρχουν σε αποκεντρωμένο επίπεδο, ούτως ώστε όταν κάποια στιγμή περατωθεί η κρίση να υπάρξει μια ανάκαμψη. Η έννοια λοιπόν του καταπιστεύματος είναι ε, συνδεδεμένο με την αρρωγή, την αποκατάσταση και την ανάπτυξη. Αυτά τα τρία πράγματα συνδέονται μεταξύ τους. Άμεση βοήθεια στον πληθυσμό, ούτως ώστε να καλύψουμε τις βασικές του ανάγκες όπως την υγεία, ε, επιστηστική ασφάλεια, ε, καταφύγια, συμφιλίωση και προσπαθούμε να φτιάξουμε λιγάκι το σύστημα, τις υπηρεσίες δηλαδή και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ε, δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2014 για μια πενταετία ε, με πρωτοβουλία της ε, Γαλλίας και αμέσως μετά η Γερμανία ε, και η Ολλανδία και ένα χρόνο μετά η Ιταλία και η Ελβετία. Ε, έχουμε και ένα κράτος που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που συμμετέχει στο καταπίστευμα. Τα καταπιστεύματα αυτά είναι ανοιχτά και σε μη ενωσιακά κράτη για να συνεισφέρουν. Όπως είπε η κυρία Μακάβεν, έχουμε 200 43 εκατομμύρια. Αν σκεφτείτε τον, τον πληθυσμό που είναι 5 εκατομμύρια, δεν είναι μικρό το ποσό αυτό ε, κατά κεφαλήν. Είναι αρκετά μεγάλο το ποσό κατά κεφαλήν. Αυτό το ποσό των δεσμεύτων, από αυτές τις δεσμεύσεις, το 98% έχει ληφθεί ήδη και έχουμε δεσμευτεί μέσω προγραμμάτων, το, έχουμε δεσμεύσει το 82%. Έχουμε συμβάσεις για το 92% και έχουμε πληρώσει πάνω από το 67% των ποσών. Ε, η δυνατότητα δηλαδή απορρόφησης υπάρχει. Ε, ήμασταν αρκετά γρήγοροι για να αποφασίσουμε για δράσεις και η εστίαση των δράσεων, εκεί που παρεμβήκαμε, εφαρμόσαμε τα προγράμματα. Φυσικά είναι δύσκολη η εφαρμογή σε μια χώρα όπως η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, γιατί υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας. Ε, χρησιμοποιούμε μη, διεθνής όσο μπορούμε περισσότερο, προσπαθούμε να ενσωματώσουμε και κάποιες τοπικές ΜΚΟ ε, για να ενισχύσουμε το δυναμικό τους, ε, φυσικά διεθνείς υπηρεσίες του ΟΗΕ, αλλά και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού παρεμβαίνουμε τώρα. Θα δείτε ότι πάνω από 40% από αυτά που κάνουμε στον τομέα της υγείας. Είναι η βασική υπηρεσία που προσπαθούμε να καλύψουμε. Καλύπτουμε σχεδόν, σχεδόν όλη τη χώρα. Καλύπτουμε πάνω από 2 εκατομμύρια ανθρώπους από τα 5 εκατομμύρια του συνολικού πληθυσμού σε ό,τι αφορά την υγεία. Εστιάζουμε στα παιδιά κάτω από των 5 ετών, σε γυναίκες φυσικά, εγγύους, μεγάλο κομμάτι αυτό. Και η άλλη βασική υπηρεσία είναι η ανάπτυξη της υπαίθρου, η συμφιλίωση. Υπάρχει ένα πρόγραμμα ε, και εκεί που επισκέφθηκε η κυρία Μακάβαν, εκεί παρεμβαίνουμε. Γιατί είχαμε πάρα πολλές γυναίκες θύματα που ήταν θύματα αυτής της ε, βίας λόγω πολέμου. Ε, επιστροφή του κόσμου στις αιστείες του. Ε, θα τον κόσμο που είχε εκτοπιστεί. Ε, υπάρχουν και πρόσφυγες εκτός της χώρας για να επιστρέψουν στην περιοχή, αλλά για να μπορέσουν να επιστρέψουν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. να υπάρχουν γεωργικά προϊόντα, θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια συστήματα συμφιλίωσης το, του λαού. Αυτά τα 4-5 χρόνια λοιπόν που δραστηριοποιούμαστε, οργανώσαμε, οργανωθήκαμε, μάλλον οργανώσαμε μια μεγάλη διάσκεψη δωρητών τον Νοέμβριο του 2016 με παρουσία και του Κοινοβουλίου. Η Λίντα Μακάβαν ήταν παρούσα. Και ελπίζουμε με την δημοκρατική μετάβαση το 2016, με τον νέο πρόεδρο που εξελέγει, η χώρα θα έμπαινε σε μια καλύτερη κατάσταση. Συγκεντρώσαμε 2 δισεκατομμύρια για αυτά τα τρία πρώτα χρόνια για ένα εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Το 2017 και το 2018 η κατάσταση όμως δεν βελτιώθηκε, επιδεινώθηκε μάλιστα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια ε, που ήταν άθλια. Είχαμε 14-15 ένοπλες ομάδες που έλεγχαν το 80% του εδάφου της χώρας. Επομένως, Φυσικά είμαστε εκεί με την αποστολή κατάρτισης ε, του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου για να στηρίξουμε τις ε, στρατιωτικές δυνάμεις, ε, τι ανώπλε δυνάμει, δηλαδή, αλλά και στην τομέα τη δικαιοσύνη και τη αστυνομία προσπαθήσαμε να συνεισφέρουμε. Τον Οκτώβριο πέρυσι με τα κράτη-μέλη και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σκεφτήκαμε τι πετύχαμε. Έχουμε πετύχει τη δυνατότητα ο πληθυσμό να έχει πρόσβαση σε βασικέ υπηρεσίε, ε, να αντέξει την κατάσταση. Αλλά υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να συνεχίσει να, βελτι... λειτουργεί το καταπίστευμα. Δεν βελτιώνεται η κατάσταση και η Νευτική Συμφωνία ε, έχει καθυστερήσει. Σε καμία περίπτωση δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει βελτιωθεί η ασφάλεια στη χώρα. Επομένως, τι έφερε το καταπίστευμα αυτό, όπως είπα πριν, ευελιξία, Δρούμε γρήγορα, προσαρμοζόμαστε, χάρη σε αυτό αλλάξαμε μερικές φορές ε, και τι περιοχέ που δραστηριοποιούμαστε λόγω προβλημάτων ασφάλειας. Ε, μπορούμε να αλλάξουμε γρήγορα το, τον τόπο δράση. πάμε αλλού. Ε, είχαμε επαφή με τι αρχές, ε, έχουμε και ένα εκπρόσωπο από την πρεσβεία. Οι αρχές μας βοηθάνε, είναι τμήμα του του Στρατηγικού Συμβουλίου και συναποφασίζουμε για τα πώς, το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια. Υπάρχει λοιπόν ένα ενωσιακό εργαλείο, το αναγνωρίζουν όλοι, το ξέρουν όλοι, όπου και να πάμε, ο κόσμος ξέρει τον Μπεκού, ε, το Ταμείο. Αυτό πρέπει να συνεχίσουμε. Το Στρατηγικό Συμβούλιο, λοιπόν, ε, έλαβε χώρα στον ε, και ζήτησε επίσημα μία παράταση. Εμείς προτείναμε μία παράταση μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020. Στα πλαίσια δι' αυτού του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Δηλαδή δεν θα πάμε στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Μέχρι το 2020 θα φτάσουμε μόνο. Θα μα επιτρέψει να καταναλώσουμε τα, να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια που έχουμε. Έχουμε υποσχέσει για επιπλέον συνεισφορέ από τη Γαλλία, κυρίω τη Γερμανία και την Ιταλία και την Ελβετία, εσχάτω, ε, συν ε, κάποια κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλά τα κονδύλια και επιπλέον έχουμε την Ειρηνευτική Συμφωνία που υπογράφηκε το Φεβρουάριο στο Παγκή μετά από κάποιες συζητήσεις ε, στο Καρτούν υπό την αιγίδα της Αφρικανικής Ένωσης. Ε, ήταν πολύ σημαντικό όταν ε, επικεφαλής η Αφρικανική Ένωση και συμφωνία με την δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση και τον πρόεδρό της. Έχουμε λοιπόν αυτή την ειρηνευτική συμφωνία που υπέγραψαν όλες οι ενόπλες ομάδες και είναι τώρα η ευκαιρία για να ξαναμπεί σε τροχιά η χώρα, να βγει από την κρίση και το Μπεκού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα ευέλικτο εργαλείο που θα υποστηρίξει την Ευτική Συμφωνία, που θα, επιστρέψει, που θα βοηθήσει τους ανθρώπους που επιστρέφουν στις αιστείες τους και δεν μπορούσαν πριν. Ε, και τώρα μπορούμε να, να παρεύουμε σε αυτές τις περιοχές. Πριν δεν μπορούσαμε λόγω της έλλειψης ασφάλειας. Ε, η κυβέρνηση όμως χάρη σε αυτό θα μπορούσε, ε, μπορεί και να στηρίξει την ενευτική διαδικασία. Τελευταία πληροφορία, πήγαμε στο Συμβούλιο, στην ομάδα εργασίας Κοντεύ, στις 14 Φεβρουαρίου και είχαμε αντίστοιχη διαδικασία, δηλαδή το Συμβούλιο Κοινωνικών Θεμάτων και Προστασία του Καναλωτή ενέκρινε την επιστολή. Έχουμε μια επιστολή από τον πρόεδρο του Συμβουλίου προς τον Επίτροπο Μίμητσα που δίνουν το πράσινο φως για την παράταση. Αυτό προς ενημέρωσή σας. Νομίζω ότι μπορώ να σταματήσω εδώ και να μου υποβάλλετε ερωτήσεις. Πριν δώσω το λόγο και πάλι στον κύριο Αρτουή για τις ερωταπαντήσεις, έχουμε εδώ τον κύριο Μάριο Σεντεζίου, ο οποίος είναι από την πρεσβεία της Κεντροαφρικανικής ε, Ένωση. Οπότε, δημοκρατία, συγγνώμη. Οπότε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που δίνετε την ευκαιρία και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία να έρθει και να απευθυνθεί στο σώμα σας. Κύριε Πρόεδρε, το Μπεκού είναι η Ευρώπη. Είναι η Ευρώπη, η γενοδορία της, είναι η Ευρώπη, οι αρχές της, η ειρήνη, η αντοχή, όπως επίσης και η ανάπτυξη η οποία θα είναι χωρίς αποκλεισμούς. Σήμερα λοιπόν η κεντροαφρικανική δημοκρατία ταυτίζεται με τον Μπεκού και στις συζητήσεις στρατηγικού περιεχομένου που έλαβαν χώρα τον Οκτώβριο εδώ στις Βρυξέλλες ε, με εξέπληξε ο υπεύθυνο του οικονομικού σχεδιασμού που είπε ότι δεν πρόκειται μόνο για υλική τεχνική στήριξη, είπε τι αντιπροσωπεύει τον Μπεκού για την περιοχή μας. Έχει ευελιξία, οπότε προσαρμόζεται κάλλιστα στην ε, παγίωση της ειρήνης. Σχέδιο της κυβέρνησης με τους εταίρους της. τον Μπεκού δρά λοιπόν στις συνιστώσεις του σχεδιασμού αυτού και έτσι σήμερα μπορούν οι κεντροαφρικανοί να σχεδιάσουν ένα καλύτερο μέλλον για τους αυτούς τους. Μιλήσαμε πριν και για μικρά προγράμματα. Εμείς είμαστε πεπισμένοι, ακόμα και αν είναι μικρές οι δράσεις του Μπεκού, εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι αυτές οι δράσεις αποφέρουν τεράστιους καρπούς. Και πιστεύουμε ότι στο μέλλον θα έχουμε ακόμα ε, μεγαλύτερα αποτελέσματα. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια ευκαιρία στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Είναι ειρηνευτικέ συμφωνίες ε, που υπογράφηκαν στις 6 Φεβρουαρίου. Ακόμα υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν έχουν γίνει καλά κατανοητά για τι συμφωνίε αυτέ, αλλά πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε αφιβολία θα διαλυθεί πολύ σύντομα. Οπότε έτσι το Μπεκού μπορεί να δράσει ακόμα πιο αποτελεσματικά. Γιατί μέχρι σήμερα ε, ξέρουμε ότι υπάρχει κάποια ανασφάλεια, κάποια βεβαιότητα, ε, το Μπεκού δεν μπορούσε να φτάσει σε κάποιες περιοχές της χώρας, ενώ τώρα με τις ειρηνευτικές αυτές συμφωνίες το Μπεκού μπορεί να κάνει περισσότερα, μπορεί να προχωρήσει περισσότερο στη δράση του και να επιτρέψει στους νέους της ε, Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, στις γυναίκες, να ελπίσουν για ένα καλύτερο μέλλον. Οπότε εμείς εδώ επιβεβαιώνουμε την βούλησή μας για παράταση του ταμείου αυτού. Και επίσης θέλουμε να πούμε ότι εσείς, εκτός από ευρωβουλευτές, εκπροσωπείτε και τις χώρες σας. Και εμείς θέλουμε να κάνουμε έκκληση σε εσά προκειμένου εσείς να εκπροσωπήσετε τη φωνή της κεντροφρικανικής δημοκρατίας στις χώρες σας, ώστε να συνεισφέρουν ε, και αυτές στο Ταμείο Μπεκού. Γιατί πρόκειται για ένα σύνολο το Μπεκού, το Ταμείο Μπεκού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της και με αμοιβαία κατανόηση μπορεί να βοηθήσει την υλοποίηση αυτού του ιδεόδους που είναι η ειρήνη και της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό είναι το μήνυμα που ήρθαμε να σας μεταφέρουμε εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος κύριε Μακάβεν. Συμφωνώ σίγουρα ε, μαζί σας που λέτε ότι το Ταμείο Μπεκού για τη χώρα σας είναι η σχέση της χώρας σας με την Ευρώπη. Το ξέρω, ναι, το καταλαβαίνω. Ε, μου είχαν φτιάξει ένα καπέλο δεν είχα πάει εκεί πέρα που το έλεγε αυτό σαν ε, μήνυμα. Οπότε θα ήταν πολύ κρίμα να σταματήσει αυτό το ταμείο. Τώρα θα περάσω το λόγο πάλι στον πρόεδρο Αρτουή που θα διευθύνει τη συνέχεια των εργασιών. Κύριο Αρτουή, πάρα πολλά επιχειρήματα, πολύ πιστικά, πράγματι, για να παραταθεί η ζωή και η λειτουργία αυτού του Ταμείου Μπεκού. Δεν ε, ξέρω αν έχει ζητήσει κανείς εδώ το λόγο. Οι συνάδελφοι. Α, εσείς, παρακαλώ, η κυρία Κέγκε. Ευχαριστώ. Σας δίνω λίγο χρόνο, να βάλετε τα ακουστικά σας. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση, που ήταν πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ τη Λίντα, που μας έδωσε όλα τα στοιχεία, που είναι πολύ σημαντικά, ότι μας είπε ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτό το ταμείο, αλλά χάρη σε αυτό και μέσω αυτού να στηρίξουμε και την ε, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Την ξέρουμε πάρα πολύ καλά την κατάσταση, την ξέρουμε στην ΤΕΒΕ. Υπάρχει και ένα άλλο πρόγραμμα που έχουμε εξετάσει την ομάδα εργασίας που αφορά τη συμφιλίωση και την ειρήνη στη χώρα αυτή για να βοηθήσουμε τον πληθυσμό της μέσω της ειρηνευτικής διαδικασίας να περάσει σε μια φάση ανάπτυξης. Και εγώ στηρίζω αυτό το καταπιστευματικό ταμείο. Πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει στην παγίωση της ειρήνης σε μια χώρα που ζει σε πόλεμο ε, εδώ και χρόνια. Τα πρώτα θύματα είναι οι γυναίκε και παιδιά. Στηρίζω και την ειρηνευτική διαδικασία, γιατί χωρί ε, ειρήνη δεν υπάρχει ανάπτυξη. Αν καταφέρουμε να του δώσουμε την ευκαιρία να παρατείνουν αυτό το ταμείο, θα υπάρξουν θετικέ απαντήσει. Εμείς έχουμε ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια να του στηρίζουμε και δεν μπορούμε να σταματήσουμε στα μέσα τη πορεία. Πρέπει να πάμε στο τέλο. Οι γυναίκε και τα παιδιά που είναι τα πρώτα θύματα χρειάζονται στήριξη. Ακόμα και μέσω αυτών των μικρών προγραμμάτων ε, για τα οποία μιλήσατε πριν. Εγώ δεν πήγα ε, μαζί με τη Λίντα στην επίσκεψη αυτή, αλλά το θέμα το ξέρω αυτό. Ε, ξέρω πολύ καλά και έχω έρθει σε επαφή με τις αρχές ε, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. Ε, συνομιλούμε στην ε, κοινοβουλευτική συνέλευση ΑΚΕ Καραϊβικής Ειρηνικού. Ευχαριστώ την Κομισιόν για τα λόγια που είπε, για αυτό που μας είπε και μέσω της γραπτής επιστολής. Ευχαριστώ και την Πρεσβεία, γιατί εμείς ως Ευρωβουλευτές πρέπει να παίξουμε ο καθένας ρόλο του. Πρέπει ο καθένας από εμά να προσπαθήσουμε να πιέσουμε τη χώρα μας, ούτω ώστε να μπορέσει η κεντροαφρικανική δημοκρατία να επανέλθει σε μια τροχιά ειρήνης και ανάπτυξης, που είναι απαραίτητο, απαραίτητη όχι μόνο για την χώρα αυτή, την κεντροαφρικανική δημοκρατία, αλλά για ολόκληρη την κεντρική Αφρική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Φυσικά όλοι επιθυμούμε η κεντροαφρικανική δημοκρατία να επανέλθει σε ειρήνη και σε ρυθμό ανάπτυξης που γεννά ελπίδα και εμπιστοσύνη για όλους τους κατοίκους. Και τώρα, θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα μεθοδολογικού χαρακτήρα. Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Προϋπολογισμών κυρίως επιθυμούν να υπάρχει ενότητα στον προϋπολογισμό. Ο πολλαπλασιασμός των καταπιστευμάτων όμως παραβαίνει αυτή τη βασική αρχή της δημοσιονομικής ενότητας. Γιατί μια τέτοια ενότητα θα επέτρεπε μια καλύτερη αναγνωσιμότητα, μια, έναν προϋπολογισμό πιο κατανοητό από τους πολίτες. Ε, η ενδιάμεση έκθεση υποβλήθηκε στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Έτσι, και εκεί υπενθυμίσαμε ότι θέλουμε να υπάρχει αυτή η δημοσιονομική ενότητα και εκφράσαμε την επιθυμία να υπάρξει μια τάξη σε, αυτή την, σε αυτόν τον πολλαπλασιασμό ειδικών εργαλείων και ταμείων που έχουν σαν αποτέλεσμα δημιουργείται ένας δημοσιονομικός γαλαξίας, όπως είπαμε. Ε, φανταστείτε ένα διάγραμμα όπου υπάρχει η καρδιά του συστήματος, δηλαδή ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, εν συνεχεία, διάφοροι γαλαξίες από ταμεία, ε, εργαλεία, ε, προσαρτήματα στον προϋπολογισμό και γίνεται έτσι ακατανόητος ο προϋπολογισμός τελικά. Θα ήθελα λοιπόν επί της αρχής αυτής να μας εξηγήσει η Κομισιόν και ποια είναι η προστιθέμενη αξία. Μας εξήγησε την προστιθέμενη αξία, μας είπε ότι το 2014 δημιουργήθηκε αυτό το ταμείο γιατί υπήρχε μια κατάσταση επίγουσα. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι πέντε χρόνια μετά Είμαστε πάντα σε μία αντίστοιχη επίγουσα κατάσταση. Επίσης, αν στραφούμε προς το μέλλον, αν φανταστούμε το επόμενο πολιετές πλαίσιο, θα πρέπει να διατηρήσουμε και σε αυτό τα καταπιστεύματα ή μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι απαραίτητες πιστώσεις θα εντάσσονται στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν υπάρχουν συνεισφορές από διάφορες χώρες, για να εκφράσουν την αλληλεγγύη και την γενναιοδορία τους, θα έχουμε τη δυνατότητα να προσφύγουμε στους, στις πόρου, στους δεσμευμένους πόρους, στις δεσμευμένες πιστώσεις. Η Κομισιόν θα ήθελα λοιπόν να μας διευκρινίσει ποια είναι η συμπληρωματικότητα αυτού του ταμείου σε σχέση με άλλα προγράμματα χρηματοδότησης και παρέμβασης της Ένωσης ε, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Και τέλος, θα ήθελα να ρωτήσω τη Γενική Διεύθυνση προπολογισμού να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν λάβαμε έκθεση για τα καταπιστεύματα από τον Νοέμβριο του 2018 και μετά. Έκτοτε σίγη ηχθείως από την Κομισιόν. Και μία ακόμη ερώτηση και ίσως να μπορέσετε να απαντήσετε μαζί. Σε 40 εκατομμύριο νομίζω ότι ανέρχεται το αίτημα ε, χρηματοδότησης για την παράταση του Ταμείου. Από το EDF ε, γνωρίζουμε από πού ακριβώς παίρνουμε τα χρήματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να προσπαθήσω καταρχάς να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις και η συνάδελφός μου, η Δεσποινή Νιμάρο, θα σας δώσει σίγουρα κάποια συμπληρωματικά στοιχεία. Όσον αφορά την πηγή χρηματοδότησης του Ταμείου Μπεκού, Ήδη έχουν αναφερθεί τα 243 εκατομμύρια ως το σύνολο των δεσμεύσεων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2018. Από αυτά τα 243 εκατομμύρια, τα 67 ε, αποτελούν δέσμευση άλλων χορηγών, ενώ τα τέσσερα κράτη-μέλη και η Ελβετία ήδη αναφέρθηκαν ως αυτή η άλλη χορηγή. Το τα 67 εκατομμύρια αντιπροσωπεύουν το 28% των 243 εκατομμυρίων. Το υπόλοιπο λοιπόν θα προέρχεται είτε από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 63 εκατομμύρια, 26%. Και η μεγαλύτερη μερίδα προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, συνολικά 113 εκατομμύρια, που αντιπροσωπεύει το 46%. Αυτή λοιπόν είναι η ανάλυση της χρηματοδότησης. Κύριε Αρτουή, μπορεί να υπάρχει κάποια παρανόηση. Θα ξαναελέγξω τις εκθέσεις που λογικά λαμβάνεται κάθε μήνα. Έχω εδώ μπροστά μου την ε, έκθεση της 31ης Δεκεμβρίου που από ό,τι γνωρίζω θα πρέπει να έχετε λάβει, αλλά θα το ξαναελέγξω και θα σας απαντήσω. Αλλά από ό,τι γνωρίζω, λογικά θα πρέπει να έχετε λάβει τις εκθέσεις. Μια τρίτη ερώτηση που θα μπορούσε να ε, τεθεί στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμών θα υπάρξει ανάγκη για νέα καταπιστευματικά ταμεία στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρί να απαντήσουμε σε κάτι τέτοιο. Είναι σαφέ ότι ο νέος Δημοσιονομικό Κανονισμό προβλέπει τη δυνατότητα αυτή. Είναι επίση σαφέ ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει σε οποιαδήποτε τέτοια απόφαση. Είναι επίσης σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει προτάσεις για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο Μπορεί τελικά όμως η ανάγκη για καταπιστευματικά ταμεία να είναι μικρότερη κατά τη διάρκεια του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να απαντήσουμε σήμερα σε αυτό. Εάν όμως η ευελιξία που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετηθεί, τότε μπορεί να υπάρχει λιγότερη ανάγκη για καταπιστευματικά ταμεία ε, στο επόμενο πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Δίνω το λόγο στη συνάδελφο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, τέθηκαν ε, κάποιες ερωτήσεις. Γιατί, για παράδειγμα, είναι ακόμη επίγουσα η ε, δραστηριότητά μας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Εάν κοιτάξετε τα στοιχεία για την κατάσταση του πληθυσμού, πάνω από το 50% χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια το ποσοστό εκτοπισμού είναι ε, πολύ υψηλό, το ποσοστό θνησιμότητας ε, είναι πολύ υψηλό, έχουμε πρόσφυγες ε, έξω από τη χώρα, έχουμε παιδιά που τα τελευταία χρόνια δεν έχουν πάει σχολείο, είναι πολύ υψηλό το ποσοστό των παιδιών αυτών. Αυτό που ελπίζαμε εμείς ότι θα αποτελέσει βελτίωση στην όλη κατάσταση δεν έχει υλοποιηθεί. Η η ειρηνευτική συμφωνία υπεγράφει 6 Φεβρουαρίου μόλις πριν από 1,5 μήνα, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία. Θα πρέπει να φροντίσουμε οι ένοπλες ομάδες ε, να αφοπλιστούν, να είναι διατεθειμένες ε, να ενσωματωθούν ε, σε κάποιο είδο νόμιμης ζωής, διότι η παρανομία του δίνει πολύ πιο ψηλά κέρδη. Θα πρέπει λοιπόν να του δώσουμε κίνητρα για να αφοπλιστούν και να ενταχθούν στην κοινωνία. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια δημιουργία συμφιλίωσης ανάμεσα στις διάφορες κοινότητες, διότι πολλέ από τις κοινότητες αυτές έχουν επηρεαστεί από την βία ανάμεσα στι διάφορε ομάδε. Πολλή δουλειά λοιπόν απομένει να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση. Επίσης, ε, οι δυνατότητες ε, του κράτους ε, συνδέονται με την ασφάλεια. Εάν δεν έχουμε κατάσταση ασφάλειας, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε η οικοδόμηση του κράτους. Ξεκινάμε. Σε κάποιες πόλεις είναι κάτι όμως που θα απαιτήσει χρόνο. Είναι λοιπόν μια διαδικασία την οποία θα πρέπει να παρακολουθήσουμε στενά. Ρωτήσατε το ποια είναι η συμπληρωματικότητά του με τα άλλα ταμεία και τα άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το καταπίστευμα Μπεκού ξεκίνησε το 2014, όταν δεν είχαμε τίποτα ακόμα σε διμερές επίπεδο. Δεν είχαμε δηλαδή ενδυθικό εθνικό πρόγραμμα ε, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, γιατί αυτό υπογράφηκε μόνο το 2017. Στην αρχή δράσαμε λοιπόν με κάποια ταμεία ε, και την πασαρέλα του Ευρωπαϊκού Αμυντικού, ε, Αναπτυξιακού Ταμείου με στόχευση ιδιαίτερη, ούτως ώστε να βοηθήσουμε το κράτος να αναλάβει τις βασικές του ευθύνες, να πληρώνει τους μισθούς καταρχάς. Ε, στηρίξαμε τον προϋπολογισμό για να πληρώνει ένα ελάχιστο μισθό στους υπαλλήλου, ούτως ώστε να μην καταρρεύσει το, το κράτος. Αυτό το κάναμε το καταπίστευμα λοιπόν. Και συνεχεία ε, κάναμε όλο και περισσότερα. Το 2017 ε, υπογράψαμε το Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα, ε, φτιάξαμε ένα πιο πλούσιο, ας πούμε, ε, πρόγραμμα στήριξης, ε, ούτως ώστε τα διάφορα να στηρίξουμε και την υγεία και τον κοινωνικό τομέα και να δίδονται και διάφορα ε, ποσά που πρέπει στον κόσμο. Το 2018 ασχοληθήκαμε με την μεταρρύθμιση της ασφάλειας. Ε, παρεμβαίνουμε σε επίπεδο αστυνομίας και δικαιοσύνης. Ε, συνδυάζοντας αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της άμυνας ε, μαζί με το προς, τους, ε, προς δυνάμει. δυνάμεις. Δεν έχει κανένα νόημα να ασχολούμαστε και να αναπτύσσουμε τις ένοπλες δυνάμεις αν δεν υπάρχει ποινικό σύστημα, αν δεν υπάρχει αστυνομία. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να στηρίξουμε την αστυνομία και την δικαιοσύνη, ειδικά το ποινικό κομμάτι. Ε, αυτά. Και το τελευταίο ερώτημα της κυρίας Μακάβεν για τις μελλοντικέ χρηματοδοτήσεις ήταν αυτό. Μου είπαν ότι υπάρχουν ακόμα 40 εκατομμύρια. Ναι. Από πού προέρχονται? Από το Ευρωπαϊκό Ταμείο ανάπτυξη, Από το γενικό απόθεμα? Ή από το 11ο ενδεικτικό πρόγραμμα για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Προτείναμε πέρα από αυτά που δίνουν επιπροσθέτως τα κράτη-μέλη πέρα από αυτά, από τη Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και τώρα την Ελβετία, που μπορούν να φτάσουν τα 70 εκατομμύρια όλα μαζί, προτείναμε ε, άλλα 40 εκατομμύρια από το 11ο ενδεικτικό αποθεματικό του Ταμείου Ανάπτυξης για να συμπληρώσουμε το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. Κάποια από αυτά τα λεφτά θα πάνε στον Μπεκού κατευθείαν ε, και σκεφτόμαστε όμως βεβαίω και τον επόμενο εκλογικό κύκλο. Θέλουμε να τον στηρίξουμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικός. Είναι προτεραιότητα για την Ένωση. Ίσως μπορώ να σταματήσω εδώ. Για αυτούς που δεν ε, ξέρουν ε, τα αναπτυξιακά και τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, ε, υπάρχει χρηματοδότηση της, του ανθρωπιστικού κομμάτι σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Δεν νομίζω ότι γίνεται με βάση τους κανόνες. Ε, είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο νέο μας πρόγραμμα. Ε, πρέπει να δούμε την ε, σύνδεση ανάμεσα στην ανθρωπιστική βοήθεια και την μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή βοήθεια. Ε, αυτά πρέπει να τα χρηματοδοτήσουμε. Ελπίζουμε το νέο πρόγραμμα να υπάρξει χρηματοδότηση. Μακροπρόθεσμες κρίσεις που μπορούν να έχουν χρηματοδότηση πολυετή όσοι ε, ξέρουν τα αναπτυξιακά θέματα, ξέρετε πολύ καλά τι κάνουν τα καταπιστεύματα. Το θέμα είναι μακροπρόθεσμα, πώς θα στηρίξουμε σε περίπτωση ε, πολύχρονης ανθρωπιστικής κρίσης. Μην μιλάς. Πρόεδρε, μια και κανείς δεν αμφισβητεί την ιδέα της παράτασης του Ταμείου, και η κυρία Κιέγγι που μίλησε ήταν υπέρ. Επομένως θα μπορούσα να ετοιμάσω τα απαραίτητα έγγραφα για τους ε, συντονιστές για να ετοιμάσουμε την επιστολή προς τον Ταγιάννη. Για να στηρίξουμε και εμείς την παράταση του Ταμείου. Και το άλλο το θέμα που θέσατε για την ενότητα του προπολογισμού, να υπάρχει ένας ενιαίος προπολογισμό, συμφωνώ βεβαίως. Κάποια στιγμή μου δείξατε ε, το σχέδιο με όλε τι διάφορε χρηματοδοτήσει που είναι διασκορπισμένε. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να πλουστευτεί αυτό το σχέδιο. Αλλά αυτό θα πρέπει να το κάνει επιπλέον, μάλλον, το επόμενο δημοσιονομικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για το παρόν δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι το 2020. Συμφωνούμε λοιπόν με την παράταση, στηρίζουμε αυτή τη νεαρή δημοκρατία που χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει άλλους εταίρους αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ <clears throat> απόλυτα με το συμπέρασμά σας. Έτσι όπως το διατυπώσατε αγαπητή Λίντα. Το υπενθύμησε και ο συνάδελφος ότι πρέπει να υπάρχει ευελιξία αν θέλουμε τη διατήρηση των καταπιστευματικών ταμείων στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί δημιουργούμε πολλά καταπιστευματικά ταμεία επειδή είναι άκαμπτο το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και δεν υπάρχει αρκετό περιθώριο ευελιξίας. Οπότε το μήνυμα νομίζω ότι εισακούεται. Τώρα, τυπικά, για να έχουμε ένα σχέδιο βοήθειας που θα στείλουμε με γραπτή διαδικασία στους συντονιστές των επιτροπών μας, και όταν θα έχουμε καταλήξει την επιστολή θα τη στείλουμε στον πρόεδρο Ταγιάννη και θα υπάρξει και ανακοίνωση στην Ολομέλεια την επόμενη ή την τελευταία αυτής της θητείας, του Απριλίου δηλαδή, και υπό αυτές τις συνθήκες πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να επιτρέψουμε στο Ταμείο να λειτουργήσει 18 ακόμα μήνες μετά την εκπνοή του. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την κοινή συνεδρίαση που είχαμε οι δύο επιτροπές μας μαζί. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Λίντα, ευχαριστώ και τους συναδέρφους της Επιτροπής Ανάπτυξης. Θέλω να πω στους συναδέρφους της ΔΕΒΕ ότι έχουμε και με την Ίντεκο Επιτροπή τώρα κοινή συνεδρίαση. Και σας, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ γενικά για την συνεργασία σας όλα αυτά τα πέντε χρόνια, όχι μόνο για τη σημερινή συνεδρία. Η δικιά σας Επιτροπή πάντα στήριζε την ανθρωπιστική και την αναπτυξιακή βοήθεια. Η βοήθειά σας ήταν πολύτιμη.